Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε γρήγορα. Ίσως θα καταφέρουμε μάλιστα να τελειώσουμε και λίγο νωρίτερα. Θα το χαλάσω στο τέλος αυτό με το σφυρί μου. Μ' αρέσει αυτό το σφυράκι. Nein, das tue ich nicht. Nein, ich schmeiße nicht mit Hammern um mich. Λοιπόν, συνάδελφοι, αν ξεκινήσω νωρί, θα τελειώσω νωρί. Λέω να προχωρήσουμε για να μην χρειαστεί να τρέχουμε στο τέλος και να περάσουμε στο σημείο 9, προϋπολογισμός 2018, γνωμοδότηση, εντολή για τον τριημερή διάλογο. Ο κ. Μόρτεν Λόκεγκαρντ είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης από πλευράς μας. Πολλοί είχαν και σε προηγούμενες θητείες και σε προηγούμενες χρονιές να συνεργαστούν με τον Μόρτεν σε ζητήματα προϋπολογισμού. Γι' αυτό ε, χαιρόμαστε πολύ Μόρτεν που είσαι άλλη μια φορά εδώ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η Δευτέρα Μαΐου, αύριο, ε, πολύ σύντομα μάλλον, και η συζήτηση ε, στην ε, δική μας Επιτροπή θα γίνει ε, στις 30 Μαΐου. Καθήλυνα αρμόδια επιτροπή φυσικά είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Να δώσω το λόγο στον Μόρτεν χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ και για τα καλά εισαγωγικά σας λόγια. Είναι ωραίο να έρχομαι σε αυτή την όμορφη και σπουδαία επιτροπή. Έχω και ένα ντεζαβί μάλιστα. Αισθάνομαι ένα ντεζαβί. Όταν για πρώτη φορά ήμουνα εισηγητής, ε, ήμουν εισηγητής και στην προηγούμενη θητεία. Γι' αυτό λοιπόν το έχω ξαναδεί το έργο. Και τελευταία φορά το ευχαριστήθηκα, το διασκέδασα και νομίζω ότι και αυτή τη φορά το διασκεδάσω. Θα δούμε πάντως. Τα πάντων, χαίρομαι που είμαι εδώ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να τονίσω τα βασικά σημεία της νομοδότησης. Ακούσατε ότι βασίστηκα στα συμπεράσματα της ε, Επιτροπής σας, τα περσινά, τίποτα το καινούριο λοιπόν εδώ. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι και ισορροπημένη και να μην δημιουργεί διχογνωμίες στην Επιτροπή. Να τονίσω κάποια λίγα θέματα. Αποδοκιμάζουμε το γεγονός ότι το συμπληρωματικό κονδύλι για το πρόγραμμα Erasmus Plus ε, μειώθηκε από το Συμβούλιο ε, στα 100 εκατομμύρια Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, αν μπορούμε. Είναι από τα βασικά σημεία στη δουλειά μας. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, η προτινόμενη χρηματοδότηση για το νέο σώμα αλληλεγγύης αντλεί σημαντικούς πόρους από το Erasmus 58 εκατομμύρια συγκεκριμένα. Και το ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει μαζί, Πρόεδρε, αυτό το σημείο θα πρέπει να τεθεί ξανά. Το να παίρνεις λεφτά από το Erasmus Plus μου φαίνεται πολύ εύκολο. Μάλλον έχει πρόβλημα η Επιτροπή να βρει λεφτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα κάνω καν τη συζήτηση αν είναι καλή ιδέα ή όχι. Αν το κάνει τουλάχιστον, ε, ας το συζητήσουμε. Ας συζητήσουμε το από πού μπορεί να βρει από πού αλλού μπορεί να βρει τα λεφτά. Τρίτο σημείο. Τονίζουμε ότι και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, όσο και το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, 11 και 16% αντίστοιχα το 2016, και αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια στους ετούντες και δημιουργεί προβλήματα στην ε, λειτουργία των προγραμμάτων. Πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι στα προγράμματα το 2018, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική η λειτουργία τους. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια και αυτά τα δύο προγράμματα είναι στον πυρήνα της δουλειά μας. Θέλουμε επίσης ε, μεγαλύτερη συνέργεια ανάμεσα στα προγράμματα πολιτισμού και εκπαίδευσης, να λυθούν τα θέματα χρηματοδότησης και επιπλέον ε, να βρεθούν από την αρχή λεφτά. Να δοθούν ήδη από την αρχή λεφτά. Ε, Επίσης ε, βρέθηκαν 7 εκατομμύρια, φρέσκο χρήμα αυτό, αυτό είναι καλό. Επίσης, η νέα αφήγηση για την Ευρώπη διανύει το τελευταίο της ε, έτος. Καλό είναι να κάνουμε ένα επικοδομητικό διάλογο με την Κομισιόν για το πώς θα συνεχίσουμε αυτό το project, ούτω ώστε να ενταχθεί στα προγράμματα που θα αρχίσουν να τρέχουν από το 2020 και μετά. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, ο τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να μπορέσω μέσα στον περιορισμένο χώρο που προβλέπεται για αυτή την γνωμοδότηση να πούμε τα σημαντικά θέματα. Προσβλέπω στη συζήτηση ε, και στις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσω κι εγώ ένα θέμα που συζητήσαμε σήμερα και στις ιδρύες των συντονιστών και αναφέρομαι στο Move to Learn, Learn to Move, το πρόγραμμα αυτό που προτείνει η Κομισιόν ως πιλωτικό πρόγραμμα για αυτή την ιδέα που προήλθε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, του, Interrail, του εισιτηρίου Interrail για όλους ε, όπου και οι συντονιστές ε, σήμερα το πρωί συμφωνήσαμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε και για αυτό το σκοπό να περιοριστούν τα χρήματα του Erasmus Plus. Ε, βέβαια τα χρήματα είναι λίγα, 2,5 εκατομμύρια, αλλά 2,5 εκατομμύρια εδώ, 2,5 εκατομμύρια εκεί και κανένα 2 εκατομμυριάκια από εκεί. Ε, τελικά καταλήγουμε να έχουμε ένα εράσμου το οποίο τελικά θα χρηματοδοτεί ε, διάφορα άλλα προγράμματα. Να το τονίσουμε και αυτό. Τώρα, έχω τους σκιώδεις, τους σκιώδεις, κύριος Μαστρογεύσκη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι πολύ σπάνια ε, η κατάσταση να μπορεί κανείς να διακρίνει με τόση σαφήνεια αυτά που λέει ο συντάκτης νομοδότησης. Τρία σημεία. Μια θλιβερή διαπίστωση που δυστυχώς πρέπει να μοιραστώ μαζί σας είναι το γεγονός ότι εκ ε, γνωρίζουμε ότι πολλές φορές η Κομισιόν μας δίνει χρήματα αλλά μετά μας παίρνει και χρήματα πίσω. Είχαμε μια υπόσχεση να αυξηθούν τα κονδύλια για το Erasmus ε, Plus, το ίδιο και για τη Δημιουργική Ευρώπη. Το αποτέλεσμα όμως, ε, η αύξηση των 200 εκατομμυρίων που μας είχε υποσχεθεί κατέληξε να είναι μια αύξηση 100 εκατομμυρίων μόλις Και τώρα έχουμε πια και μια αύξηση των προγραμμάτων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από αυτά τα χρήματα. Η υλοποίηση και η εκτέλεση των, ε, των, ε, των δράσεων του Erasmus Plus είναι σημαντικό. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο και περίπλοκο είναι αυτό το θέμα, πόσο δύσκολο, και, ε, ε πόσο δύσκολο είναι στην υλοποίησή του αυτό το πρόγραμμα. Και ε, παρόλα αυτά, δυστυχώς ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το φάσμα της μείωσης του κονδυλίου. Όσον αφορά την πολιστική κληρονομιά, μια θετική είδηση, μια καλή είδηση. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετα μέσα, πρόσθετα χρήματα, ε, εν μέρη τουλάχιστον, ε, διότι ένα μέρος αυτού του προγράμματος θα ε, χρηματοδοθεί μέσω του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Στην ουσία μοιράσαμε δηλαδή, επιμερίσαμε δηλαδή εδώ ε, τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Υπάρχει και αυτή η καλή είδηση, ας την αναδείξουμε. Τρίτο ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά τη γνώμη μου ότι αυτό δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από, το, από τη δημιουργική Ευρώπη, διότι αυτό θα περιορίσει πάρα πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια για, τα, για, για τις δράσεις αυτού του προγράμματος. Δεν, δεν πρέπει να δημιουργηθούν στενοποί, δεν πρέπει να δημιουργηθούν καθυστερήσεις. Κάθε εμπόδιο στην ε, χρηματοδότηση πραγματικά είναι επώδυνη για εκείνους που ε- ελοποιούν τα προγράμματα αυτά και δεν μιλούμε ποτέ, ε, οι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων δεν είναι ποτέ ε, ε, άνθρωποι με ιδιαίτερη οικονομική άνεση, να το πω έτσι, και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα δεδομένα του ευρωπαϊκού προπολογισμού μιλούμε, να το επενθυμίσω αυτό, για μικρά ποσά σε τελική ανάλυση. Επίσης τα πιλωτικά προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς. Και όχι μόνο αυτό. Δεν προβλέπονται και νέα χρηματοδοτικά μέσα για τα, ε, χρηματοδοτικά, για τα πιλωτικά προγράμματα. Η κυρία Τζεντήλη για τον κύριο Μόργανο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είχε προβλεφθεί, αντικαθιστώ τον συναδελφό Μόργανο που έχει μια άλλη δέσμευση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ε, σε μια ψηφοφορία. Θα σας μεταφέρω λοιπόν τις σκέψεις του όσον αφορά το θέμα που συζητάμε. Πρώτα απ' όλα μου ζήτησε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση. Κατά την άποψή του είναι πολύ καλά δομημένη και στις προτεραιότητες ε, για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Πολιτισμού υπάρχει συνένεση. Οπότε τα, αυτά που θα πω ε, προβλέπονται μόνο ως προσθήκες. Ε, πρέπει να παραλάβουμε δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το Erasmus Plus, την αναγκαιότητα να ληφθεί μέρος των χρηματοδοτήσεων υπό τη δράση κλειδί 2 και να προωθηθούν οι ευκαιρίες του Εράσμους μέσω της δράσης κλειδιού 3, όπως προβλέπεται στην εκτελεστική έκθεση από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το σώμα αλληλεγγύης, ε, πρέπει να προσθεθεί ένα κείμενο που θα επικεντρώνει ακόμη περισσότερο την προσοχή στη διάκριση μεταξύ του εθελοντισμού όπως ε, ε, πρέπει να ερμηνεύεται σωστά και μεταξύ της επαγγελματικής του δεν μπορούμε να αντικαθιστούμε ποιοτικέ θέσει εργασίας με την δωρεάν εργασία εθελοντών. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, θα είναι σημαντικό η χρηματοδότηση να εγγραφεί στον προπολογισμό βάσει τη ε, επιτευχθή σα πολιτική συμφωνία. Είναι κάτι διαφορετικό από τι σημερινέ δραστηριότητε του σημερινού προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη πρέπει να γίνει προσεκτική συζήτηση και για τις πολιτιστικές και δημιουργικές, ε, ε, τους δημιουργικούς κλάδους ε, ακολουθώντας τους ίδιους στόχους βάσει διαφορετικών όμως κριτηρίων χρηματοδότησης. Το σημαντικό είναι να προωθηθεί όπου αυτό είναι δυνατό η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο προγραμμάτων ώστε να υποστηριχθεί αυτός ο τόσο κρίσιμος για την ευρωπαϊκή οικονομία ε, τομέας και για να επανεκκινηθεί η ζήτηση, η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που θα αποτελέσουν κινητήριο μηχανή ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σημείωση διευκρίνηση στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που από τη δική της ανάλυση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων ίσως δεν εκτιμά αρκετά ότι η πολιτική ε, θα, πρέ... θα, πρέπει, θα είναι περιορισμένη αν δεν συνδυαστεί με πολιτικέ υποστήριξει τη ζήτηση και κάτι γενικό. Τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού και τη εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από χρόνια υποχρηματοδότηση στην Ευρώπη. Θα μπορούσαν να βρεθούν λύσει εφόσον υπήρχε ένας μηχανισμός χρηματοδότησης μέσω πραγματικών ιδίων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με ανεξαρτησία από τις εθνικές συμμετοχές. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο ε, ε, πλαίσιο των συζητήσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Για τα διάφορα αυτά σημεία θα ε, υποβάλουμε φυσικά τροπολογίε και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί η εξαιρετική συνεργασία όπως είχαμε τα τελευταία τρία έτη. Vielen herzlichen Dank, Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ, Πέτρα. Ευχαριστώ, Μόρτεν, για τις προτάσεις του. Γενικά, συμμερίζομαι όλα όσα είπε, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση του MFF, όπου είχαμε ε, αυτή την ε, πρόθεση αύξησης ε, των κονδυλίων για το Erasmus Plus κατά 200 εκατομμύρια και μάλιστα υπήρξε και αυτή η μείωση στα 100 εκατομμύρια από τα οποία τα 50 έχουν ήδη ιδιωτεθεί το 2017. Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Πρέπει ως Επιτροπή να επιμείνουμε το νέο σώμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην χρηματοδοτηθεί από το ε, Erasmus Plus και για τη δημιουργική Ευρώπη ο προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ χαμηλός κάτι που μειώνει και τα ποσοστά επιτυχίας, αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι διότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη απήχηση όταν υποβάλλουν αιτήσει για ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερες ε, συνέργειες μεταξύ των ε, ταμείων ΕΤΣΕ και ΔΕΤ. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι αν κοιτάσουμε ε, κοιτάξουμε τις ε, εκκλήσεις για ε, μεγαλύτερη απεύθυνση και συμπερίληψη μεταναστών και προσφύγων. Να αξιοποιηθεί το Erasmus Plus δηλαδή ε, και για αυτόν τον σκοπό. Και νομίζω ότι και από άποψη προϋπολογισμού ε, πρέπει να έχουμε και αυτό στην προσοχή μας, να το πούμε δηλαδή με σαφήνεια ότι μας ενδιαφέρει και αυτός ο τομέας της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, Julie Ward. Δύο λεπτά σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, πολύ. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν ήδη. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις επενδύσεις ε, στις τέχνες και στη δημιουργικότητα, διότι αυτό σε τελική ανάλυση μας εξοικονομεί χρήματα. Όταν επενδύουμε σε καλά πολιτιστικά προγράμματα και σε πολιτιστικές ανταλλαγές, υποστηρίζουμε ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές αξίες και διασφαλίζουμε ότι οι περιφερειοποιημένες κοινότητες θα συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο της κοινωνίας και δεν θα ριζοσπαστικοποιούνται. Ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της Τουρκίας εγώ έχω επαφή με προγράμματα, οργανώσεις ε, καλλιτεχνικές στην Τουρκία, ε, ενώσεις νέων, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δεν πρέπει να τους τιμωρούμε για αυτά που κάνει η κυβέρνησή τους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη προγραμμάτων πολιτιστικής έκφρασης με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Και ξέρω ότι το Goethe Institute ε, πρόκειται να κάνει μια πρόσθετη χρηματοδότηση και αν θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς ε, ε, συνεταίροι σε αυτό, πιστεύω θα βοηθούσε πολύ την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φρέντερικ Φίμαϊρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη Κομισιόν. Θα επιθυμούσα να σας ευχαριστήσει για την πραγματική υποστήριξη που παρέχετε στα προγράμματα αυτά, που είναι τόσο σημαντικά στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας και της νεολαίας. Είναι πολύ σημαντικό για τα καλύτερα αποτελέσματα για τους φοιτητές, για τους καλλιτέχνες, για τους φοιτητές. Είναι σημαντικό, όπως είπατε, ε, και κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και των επιπλέον ε, κονδυλίων για το Erasmus Plus. Ε, Δυστυχώ όπως και εσείς, λυπόμαστε που η αρχική πρόταση τη Κομισιόν για τα 200 εκατομμύρια επιπλέον δεν ακολουθήθηκε τελικά, αλλά να είστε βέβαιοι ότι ό,τι υπήρξε θα βοηθήσει τον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης το 2017 τομεί που μερικές φορέ παρουσιάζουν αδυναμίε και που υπάρχουν με υπάρχει τεράστιο δυναμικό επιπλέον απορρόφησης. Η υποστήριξή σας ήταν καθοριστική και για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Έτος 2018. Χαιρόμαστε για τα 4 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για το 2018, ε, τα κονδύλια ε, ανάληψη υποχρεώσεων ε, παρότι ακόμα θα χρησιμοποιηθεί για το Creative Europe. Σημαντική θα είναι η συμβολή για το δημοσιονομικό έτος 2018, παρότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών έχουμε εξαιρετικό ιστορικό ε, δημοσιονομικό υπήρξε εξαιρετική απορρόφηση των κονδυλίων, έχει ξεκινήσει πολύ καλά και το 2017. Ε, έχουμε μπει σε κανονική ταχύτητα απορρόφησης τώρα. Οπότε για το 2018 η πρόταση της Κομισιόν για τα προγράμματα αυτά ε, θα είναι ένα έτος φυσιολογικής απορρόφησης θεωρούμε το 2018. Θα ζητήσουμε τα μέγιστα ποσά βάσει των ανώτων ορίων που προβλέπονται στη δημοσιονομική προοπτική όσον αφορά τις δεσμεύσεις αναλήψης υποχρεώσεων ε, ε, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών για να απαντήσω στο, για το ερώτημα του backlog, να σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει backlog αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εκαθαρίσουμε το συσσωρευμένο backlog, οπότε βρισκόμαστε σε υγιή κατάσταση. Ε, οπότε βρισκόμαστε εκεί που θέλαμε στο επίπεδο αυτό. Επιπλέον, όπως ξέρετε, τα δημοσιονομικά προφίλ των προγραμμάτων μας ε, έχουν μείνει σε backlog. Δηλαδή αυξήσεις προϋπολογισμού με τα χρόνια ε, συσσωρεύτηκαν με τα προγράμματα και θα δούμε και αύξηση των πιστώσεων ε, σιγά σιγά ε, που διαδίδεται για το Erasmus για το Creative Europe για το 2018 προτείνεται αύξηση σε σχέση με το 2017 του 9,1% για ε, το Creative Europe και 12% περίπου για το Erasmus Plus σε πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτό περιλαμβάνει και τη δημιουργία τη δημιουργία του Σώματος Αλληλεγγύης. Και τέλος, να σας μιλήσω λίγο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η, βασική, η νομική βάση, ξέρετε, βρίσκεται υπό προετοιμασία και στόχος είναι να υποβληθεί στους επιτρόπους ε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ε, κατά την έξι της εξέτασης του προπολογισμού 2018, προβλέπεται το νέο αυτό πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί εν μέρη μέσω ε, ε, Μεταφορά κονδυλίων από άλλα προγράμματα αλλά και με χρήματα που προέρχονται από τα σημερινά ε, δημοσιονομικά περιθώρια κατά τουλάχιστον 25% ε, η ανακατανομή αυτή των κονδυλίων που είχε ληφθεί από το Erasmus Plus στην πρόταση που έχουμε ανέρχεται σε 60 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Να πω ότι μάλλον δεν θα υπάρξει ε, το σώμα αλληλεγγύης δεν θα επηρεάσει το Creative Europe. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Αυτά που είπατε για το σώμα αλληλεγγύης δεν μας χαροποιούν ιδιαίτερως, να σας το πω ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι ότι ελπίζαμε τα 50 επιπλέον εκατομμύρια που θα είχαμε στη διάθεσή μας φέτος θα διατίθενταν, ε, διατίθενταν για αυτά ε, για αυτά που πράγματι αρχικώς είχαν ε, προβλεφθεί και όχι για μια νέα, βεβαίως καλή, αλλά πάντως νέα ιδέα. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και τον ε, Μάιο. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά για όσα μας είπατε. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο ξανά στον κύριο Λόκεγκαρτ και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με, τον, με τη συζήτηση με το γενικό εισηγητή μας για τον προϋπολογισμό ο οποίος είναι ήδη εδώ. Κύριος Λόκεγκαρτ, σύντομα θα σας τα πω. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Να σας υπενθυμίσω απλώς αυτό που είπε η Πρόεδρος, ε, η προθεσμή υποβολής τροπολογιών είναι η Δευτέρα Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα. 30 ε, Μαΐου θα γίνει 13 Μαΐου μάλλον θα γίνει η συζήτηση. Ε, στα μέσα του Μαΐου θα γίνει η παρουσίαση στην Επιτροπή Προπολογισμών, όπου και θα γίνει συζήτηση και για τα ζητήματα που σχετίζονται με το σώμα αλληλεγγύης και, και άλλα βεβαίω θέματα και θα συντάξουμε και γνωμοδότηση και για αυτό το θέμα, το οποίο θα συζητηθεί στον ε, Ιούνιο και θα ψηφιστεί τον, ε, στις αρχές Ιουλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και προσβλέπω στην καλή μας συνεργασία με όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μόρτεν. Εύχομαι σε σένα και στους σκιώδεις εισηγητές καλή συνεργασία και περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Εισηγητή για τον προπολογισμό 2018, τον συνάδελφο Μούρεσαν. Καλώς ήρθατε ε, στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να κάθεστε ε, εδώ μαζί μου. Αν θέλετε να καθίσετε κάτω βεβαίως ε, δεν έχω αντίρρηση. Σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες σας για τον προπολογισμό του 2018 και με την ευκαιρία αυτή θα σας, δώσουμε, θα σας παρουσιάσουμε και εμείς τις δικές μας προτεραιότητες. Ξέρω ότι αυτόν τον καιρό κάνετε έναν γύρο και επισκέπτεστε όλες τις επιτροπές. Α, θα έρθετε τελικά στο βήμα. Καλά θα κάνετε. Yeah. <laughs> Μη φοβάστε, δεν δαγκώνω. Ξέρω λοιπόν ότι επισκέπτεστε αυτή την περίοδο όλε τι επιτροπέ. Είναι σκληρό το έργο αυτό, αλλά ω γενικό εισηγητή ε, νομίζω ότι θα σα βοηθήσει, ω γενικό εισηγητή θα σα βοηθήσει αυτό. Χαίρομαι που είστε μαζί μα Να σα δώσω τώρα το λόγο για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια θα ξαναδώσω το λόγο στον δικό μα ε, εισηγητή, τον Μόρτεν Λόκεγκαρτ, προκειμένου να σα παρουσιάσει εκείνο τι δικέ μα προτεραιότητε. Κύριε Μούρε, αν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε που με δεχτήκατε σήμερα το απόγευμα. Όπως είπε και η Πρόεδρος, επισκέπτομαι όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να συζητήσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης του 2018. Γιατί όλοι μαζί στην ε, Ολομέλεια του Μαρτίου υιοθετήσαμε την έκθεσή μου για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 και έχουμε ένα πρώτο προσχέδιο, ένα πρώτο σκαρίφημα για τις βασικές προτεραιότητες του 2018. Περιμένουμε το σχέδιο προϋπολογισμού που θα ετοιμάσει η Επιτροπή τέλος Μαΐου και εν συνεχεία πολύ σημαντικό θα είναι και για την ε, και για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή θέση και να δείξουμε ενότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουν, για να έχουμε αυτή την ενότητα, ποιε είναι οι δικέ σα προτεραιότητε. Θέλω να μου πείτε πώ βλέπετε τα πράγματα καταρχά εσεί, αφού σα πω κι εγώ ε, πώ τα βλέπω εγώ, ε, να μου πείτε κι εσεί λοιπόν ποιε θέλετε να είναι οι προτεραιότητε όταν συζητήσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τώρα είναι η αφετηρία της συνεργασίας μας, του διαλόγου μας και αφού η Κομισιόν ετοιμάσει το σχέδιο προϋπολογισμού θα είναι σημαντικό να ακούσω τις απόψεις σας για να δω πού πιστεύετε ότι πρέπει να επιμείνουμε ούτω ώστε οι τομείς στους οποίους έχουμε συναρμοδιότητα να χρηματοδοτηθούν σωστά. Οι βασικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 θα πρέπει καταρχάς να είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση και δεύτερον η ασφάλεια των πολιτών. Γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένουν οι πολίτες της ε, Ευρώπης από την Ευρώπη. Καταρχάς δουλειές και μετά ασφάλεια. Τα τελευταία δύο χρόνια καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίσαμε την κρίση με τους πρόσφυγες και όλοι οι πόροι που βρήκαμε από τον προπολογισμό της Ένωσης από το Ταμείο για την διευκόλυνση για τους Τούρκους, όπου οποιοδήποτε μέσο ε, χρησιμοποιήθηκαν. Το βασικό είναι όμως να δώσει καρπούς για τους ανθρώπους της Ευρώπης. Η πρώτη προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουμε είναι ανάπτυξη, θέση απασχόλησης, ενίσχυση οικονομίας, πιο ανταγωνιστική οικονομία, πιο ελκυστική για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να επενδύσουν σε εμά, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε υποδομέ, σε καινοτομία, σε μικρομεσαίες επιχειρήσει, στην υποστήριξη τη επιχειρηματικότητα, κυρίω των νέων επιχειρηματιών. Τα προγράμματα τα οποία θέλουν να ενισχυθούν είναι το Ορίζοντα 2020 για την ε, καινοτομία, το Connecting Europe Facility για τι υποδομέ, το κόσμο, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, για, για τους ε, με, με, μικροεπιχειρηματίες κτλ. Ε, και το Εράσμους φυσικά. Καθώς και η εγγύηση για την νεολαία. Το Εράσμους έχει αποδείξει ότι είναι βιώσιμο εδώ και 30 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι από έρευνες προκύπτει ότι οι εργοδότες όταν δίνουν δουλειά κυρίως σε νέους ε, εκτιμούν την διεθνή εμπειρία. Πάνω από 30% εργοδοτών θέλουν κάτι τέτοιο σήμερα. Το να είσαι λοιπόν τμήμα του Εράσμου σημαίνει ότι εξοπλίζουμε τους νέους της Ευρώπης με την εμπειρία που χρειάζονται, ούτω ώστε να έχουν περισσότερες και καλύτερες τύχες στην αγορά εργασίας. Το καλό για το Εράσμους είναι ότι έχουμε λάβει στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ως συνέπεια της αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου μια δέσμευση για επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος ε, του, αυτής της θητείας του 2020. Και θα πρέπει να ξέρετε ποιε είναι οι τελευταίε εξελίξει. Εμείς στο Κοινοβούλιο κάναμε ό,τι μπορούσαμε και υιοθετήσαμε όλα αυτά που έπρεπε να υιοθετήσουμε για την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Στο θεματολόγιο του Συμβουλίου, ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ήταν το θέμα αυτό σήμερα και αφού το ζήτησε το Ηνωμένο Βασίλειο, το θέμα βγήκε από την ατζέντα του Συμβουλίου. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να ψηφίσει για την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι να γίνουν οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το να το καθυστερήσουμε κατά δύο ή τρεις μήνες δεν είναι πρόβλημα. Γιατί τελικά τα λεφτά τα οποία τα υποσχεθήκαμε για, τον, ε, για το Connecting Europe Facility, για το Horizon 2020, για την εγγύηση για την νεολαία, ε, θα δοθούν, ακόμα και αν καθυστερήσουμε δύο μήνες. Αλλά... Αλλά όμως ε, υπάρχουν άλλα προβλήματα ε, για πολλά προγράμματα, για τους νέους, για την εκπαίδευση και είναι προς ε, το κοινό συμφέρον να πούμε στο Συμβούλιο μέσω όλων των διάβλων που έχουμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις του. Και η Επιτροπή σας φυσικά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την πρωτοβουλία για την νεολαία και για το Εράσμους. Για τα συγκεκριμένα προγράμματα τώρα, στον τομέα του πολιτισμού και της ηθαγένεια, φυσικά θα πρέπει να υπάρξει σωστή δέουσα προσοχή. Ένα project το οποίο έχω στο μυαλό μου, Πρόεδρε, είναι το, τα πανευρωπαϊκά δίκτυα. Κάθε χρόνο στην Επιτροπή ε, ε ασχολούμαστε με το Euronet Plus. Πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμη προβλέψιμη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει στη βιωσιμότητα αυτού του προγράμματο. Αν ναι, θα πρέπει να υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση, ούτω ώστε να μπορέσει να υπάρξει προγραμματισμό. Ε, έτσι κάνει κάθε βιώσιμος οργανισμός. Αν πιστεύουμε ότι δεν είναι βιώσιμο, τότε θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση. Και περιμένω την ε, αποψήσε το Euronet Plus. Πάντως οι διαθέσιμοι πόροι ε, υπό την επικεφαλίδα 3 είναι περιορισμένοι. Οτιδήποτε ξοδεύουμε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το ξοδεύουμε καλά. Επίσης, ξέρω και τις ε, προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Euronews ε, με την Ουκρανική εκδοχή αλλά και στην Τουρκία. Γιατί σταμάτησε η υποστήριξη από τη δημόσια τουρκική τηλεόραση, χρηματοδότηση δηλαδή, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του δικτύου, του Euronews, και εδώ η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μένα, για το πώς θα αξιολογήσουμε το Euronews σε αυτή τη φάση. Και τι οδηγίες έχετε να μου δώσετε για το Euronews και το προπολογισμό της Ένωσης. Ε, επίσης, το Ευρωπαϊκό Σώμα το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το 2018. Η πάγια άποψη του Κοινοβουλίου είναι ότι νέε προτεραιότητε θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω νέου φρέσκου χρήματο μέχρι των νέων πόρων, γιατί όταν, συμφωνούμε, ε, όταν συμφωνήσαμε για αυτό το πολιτεύσιο νομικό πλαίσιο το 2014, είχαμε κάποιε προτεραιότητε. Αλλά δεν είχαμε προβλέψει, πούμε, την κρίση των προσφύγων. Δεν είχαμε προβλέψει μέσα από τι προκλήσει του τομέα τη τρομοκρατία και τη ασφάλεια. Είναι σαφέ, λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Αν ο λαό, ε, οι κυβερνήσει περιμένουν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε και περισσότερου οικονομικού πόρου. Αλλιώ ε, τα τρέχοντα προγράμματα κινδυνεύουν. Παράδειγμα, ε, στον ορίζοντα 2020, ε, το μεγάλο project για την κοινοτομία είχε ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή τα project, τα πλαίσια του προγράμματος που μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε τα δύο πρώτα χρόνια, ε, ήταν ε, από 13% στο 9%. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά προγράμματα, project καλύτερα, που δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε πια. Και αυτό επηρεάζει φυσικά και τους νέους ερευνητέ και πολύ συχνά τις γυναίκες ερευνήτριε. Το, το ορίζοντας 2020 επηρεάστηκε γιατί ε, στον ορίζοντα 2020 και στο Connecting Europe Facility έγιναν κάποιες περικοπές όταν δρομολογήσαμε το ΕΦΣΙ, το, το, το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, όλα αυτά είναι καλά κτλ. Αλλά θα θα πρέπει να πιέσουμε σε αυτήν την περίπτωση το Συμβούλιο να δώσει νέου πόρου. Γιατί όταν βάζουμε νέα προγράμματα, θα πρέπει να βρίσκουμε νέο χρήμα για να μην επηρεάζονται τα παλιά προγράμματα. Επίση, ε, για την πρωτοβουλία για του νέου, υπάρχει μια ε, δέσμευση για να αυξήσουμε ε, κατά 1,2 επιπλέον δισεκατομμύρια μέχρι το τέλο του 2020 τη χρηματοδότηση. Από αυτά τα 1,2 δισεκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια θα πρέπει να δοθούν φέτο, το 2017. Είναι σημαντικό, όπω είπα, η αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου να περάσει, γιατί τα νέα από το Συμβούλιο είναι ε, κακά. Θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο για να υλοποιήσει τους στόχους του. Για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα σα το πω έξω από τα δόντια. Εγώ την υποστήριζα από την αρχή. Πιστεύω ότι η ανεργία των νέων είναι μία από τι βασικέ προκλήσει. Θα πρέπει να μειωθεί. Επίση, υποστηρίζω ε, αυτά τα 1,2 δι να δοθούν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα project, τα έργα δίνουν και τα αποτελέσματα που περιμένει ο κόσμος. Γιατί για μας στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι πάντα δύσκολο να δίνουμε πόρους εάν ε, λέει μια έκθεση ας πούμε ότι κάποια project, ότι κάποια έργα ας πούμε δεν είναι καλά ή τα λεφτά δεν φτάνουν στους δικαιούχους ή τα αποτελέσματα είναι φτωχά, πενιχρά. Επομένως, ναι, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, αλλά όμως αν ακούσω απόψεις και εδώ οι δικέ απόψει επίση είναι πολύ σημαντικέ. Αν φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να τροποποιήσουμε αυτή την ιστορία, να την αναθεωρήσουμε, να τη βελτιώσουμε, είμαι ανοιχτό. Γιατί τελικά θέλω να πάω στον κόσμο και να πω χρηματοδοτούμε ένα project το οποίο λειτουργεί όμω. Καταληκτικά, Πρόεδρε, τα πιλωτικά προγράμματα ή προπαρασκευαστικές δράσει. Όσο λιγότερα ε, πιλωτικά προγράμματα υποβάλλεται, τόσο καλύτερα είναι για μένα, πιο εύκολη επιλογή. Αν και θέλω πολλά πιλωτικά προγράμματα, καλά, πιστικά, πιλωτικά προγράμματα. Η διαδικασία είναι η ίδια με πέρυσι. Κάθε πιλωτικό πρόγραμμα και προπαρασκευαστική δράση πρέπει να υποβληθεί για προαξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η προθεσμία για εσάς για αποστολή των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων για προαξιολόγηση είναι η 3 Μαΐου πρέπει να στείλετε για αξιολόγηση και προγράμματα τα οποία εστάλησαν πέρυσι και τα οποία εγκρίθηκαν, αλλά τα οποία θέλετε να συνεχιστούν φέτος. Ό,τι θέλετε λοιπόν να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των πιλωτικών έργων και προσφαρασκευτικών δράσεων πρέπει να το στείλετε για προαξιολόγηση στην Επιτροπή και μετά θα φτιάξουμε ένα πακέτο το φθινόπωρο και θα δώσουμε φυσικά προτεραιότητα στα πιλωτικά έργα που έλαβαν ε, βαθμό Α από την Επιτροπή και αναμένω ότι θα μπορέσουμε επίσης να χρηματοδοτήσουμε τα πιλωτικά έργα που έχουν λάβει ε, βαθμό Β, αλλά όχι όσα έλαβαν βαθμό μικρότερο από τον Β. Οπότε πρέπει να τα στείλετε μέχρι την προθεσμία της 3ης Μαΐου οπωσδήποτε και επίσης να υπάρχει ε, σημαντικό να λάβετε και καλό βαθμό από την Κομισιόν. Αυτά από πλευρά μου, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Αναμένω τη συζήτησή μα, να ακούσω τα σχόλιά σα και ε, προσβλέπω και στη συνεργασία μα σε όλο το έτο ε, φέτο στο πλαίσιο τη εξέταση του προπολογισμού τη Ένωση. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ολοκληρωμένη οπτική που μας δώσατε σχετικά με τις προτεραιότητες σας. Νομίζω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι το Erasmus Plus βρίσκεται πάνω-πάνω στις προτεραιότητες σας. Ε, είναι πολύ θετική η είδηση αυτή. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και ιδίω μας χαροποιεί ή εμένα τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και άλλους συναδέλφους, μας χαροποιεί το γεγονός ότι το Euronet Plus ε, βρίσκεται στην ατζέντα σας Φέτος είχαμε ήδη το πρόβλημα το ότι υπήρξαν δυσκολίες διότι η Κομισιόν ε, δεν πολύ ήθελε να συνεχίσει τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες λοιπόν. Αν τα καταφέρουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε γραμμή του προπολογισμού με εξασφαλισμένο μέλλον για το Euronet Plus αυτό θα είναι πραγματικά ε, κάτι που θα ε, προσφέρει μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, γιατί νομίζω το έργο που επιτελεί το Euronet Plus είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το Euronet, είχαμε ε, πριν από λίγο μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και με προσκεκλημένους, εδώ μια δημόσια ακρόαση. Θέσαμε πάρα πολλά ερωτήματα και κατά τη γνώμη μου τα ερωτήματα δεν απαντήθηκαν ικανοποιητικά. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένω είναι και πολύ πρόημο το να ε, καταλήξουμε σε μια κοινή θέση της Επιτροπής Πολιτισμού ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή το Euronews. σε κάθε περίπτωση εκφράζονται σοβαρότατες ε, ανησυχίες τόσο ως προς την δομή του Euronews όσο και ως προς την συντακτική ανεξαρτησία, τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία. Δεν μπορώ να πω με, την, ε, με το χέρι στην καρδιά ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν όπως ε, ε, ε, ήταν μέχρι στιγμής, ούτε ως προς τη χρηματοδότηση βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού για αυτό το θέμα. Η, τα νέα από το Συμβούλιο δυστυχώς δεν είναι θετικά. Πιεστήκαμε χρονικά να εγκρίνουμε στην ουσία αυτά που ήδη έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Ε, δυστυχώς για άλλη μια φορά το Συμβούλιο και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκείνοι που πατούν το φρένο ε, αυτή τη στιγμή στο έργο μας. Ελπίζουμε σύντομα μετά τις ε, Βρετανικές εκλογές το Συμβούλιο να καταλήξει σε συγκεκριμένη απόφαση, διότι διαφορετικά ε, φοβούμε ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένα προγράμματα, κάτι που ούτε μπορούμε να αποδεχτούμε ούτε και επιθυμούμε βεβαίως. Ο Μόρτεν Λόκεγκαρ τώρα θα τοποθετηθεί και θα σας παρουσιάσει τις δικές μας προτεραιότητες και ε, μετά θα ανοίξω το λόγο για συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Να μην επαναλάβω αυτά που ήδη έχω πει. Διέτρεξα ε, ε, λίγο τις προτεραιότητες μας πέντε λεπτά πριν, ε, πριν έρθω. Να συνοψίσω πάντως λέγοντας ότι συμφωνούμε με τα περισσότερα από όσα είπε ο κύριος Μουρεσάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, αυτή την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση που μας κάνατε. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες σας ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας, τη επιτροπή Πολιτισμού. Ε, νομίζω ότι συμβαδίζουμε. Ε, βεβαίως μας ανισχύει το γεγονός ε, ε ότι μειώθηκε ο προπολογισμό του Εράσμου από το Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά, ε, είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με συγκεκριμένε προτεραιότητε για το Erasmus Plus. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο σημαντικό πρόγραμμα ε, που ε, έχει παρακολουθήσει ποτέ αυτή η Επιτροπή και στο πλαίσιο των ε, συζητήσεων για το MFF όπου είχε υπάρξει μια σημαντική αύξηση νομίζω ότι οφείλαμε να δώσουμε μια συνέχεια και νομίζω ότι αυτό θα είναι και κάτι που θα, θα κρίνει και το έργο και την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου. Επίσης θέλω να σχολιάσω το Euronet. Να πω κάτι για, την, για τη συζήτηση αυτή. Συμμετείχα πριν από ε, λίγο καιρό στην, ε, στη σχετική συζήτηση. Συμμετείχα και στην αντίστοιχη συζήτηση που είχε γίνει πριν από 5-6-7 ε, χρόνια. Η συζήτηση για το Euronet είναι, το ίδιο με, που, που γίνεται, είναι η ίδια με, με αυτή που γίνεται για το Euronews. Η γνώμη μου είναι η ίδια. Νομίζω ότι το Euronet είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, είναι ένα εξαιρετικό project ε, βρίσκεται σε, ε, σε στάδιο υλοποίηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλέ μελέτες και έχουν καταλέξει όλες στα, στα πολύ θετικά αποτελέσματα που αποφέρει. Υπήρξαν κάποιες χρηματοδοτικές δυσκολίες που οφείλονται δυστυχώ πρέπει να το πω στην Κομισιόν. Η Κομισιόν δυστυχώ, ε, ήταν πάντοτε αντίθετη με το Euronet εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Το θετικό πάντως είναι ότι οι δικέ μου πηγές λένε ότι υπάρχει μια μεταστροφή στη στάση τη Κομισιόν. Φαίνεται ότι η Κομισιόν πλέον έχει χαράξει ένα διαφορετικό δρόμο και για πρώτη φορά προωθεί μάλιστα το project αυτό, το Euronet, ε, ελπίζω να ατενίζουμε ένα λαμπρό μέλλον, ιδίω δε αν εξασφαλίσουμε και μια γραμμή του προπολογισμού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξάρουμε το έργο των ανθρώπων του Euronet με έναν, που, που το έχουν επιτελέσει με ένα πάρα πολύ μικρό προπολογισμό. Και συμφωνώ με την ανάλυση και τα συμπεράσματά σα. Πρέπει πλέον να υιοθετήσουμε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση και να λάβουμε επιτέλου μια απόφαση, η οποία για μένα είναι σαφή το ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση να προωθηθεί. Επίσης, δεν θέλω να σας κουράσω με ιστορικά δεδομένα, αλλά το Euronews έχει μια μακρά διαδρομή, ιστορική πλέον. Εγώ δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην ε, ε ακρόαση που έγινε, αλλά θέλω να... Με, ενδιαφέρει και εμένα αυτό το θέμα του Euronews, γιατί πραγματικά έχουμε χρηματοδοτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, το, Euronews, το Euronews με πολλά χρήματα, χωρίς να θέτουμε τα δέοντα ερωτήματα. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Αυτά νομίζω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος ευρωβουλευτής που θα ήθελε το λόγο ο κύριος Στογιάς και στη συνέχεια η κυρία Χέλγα Τρούπη. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Θεωρώ θετική την ευαισθητοποίηση που ακούω. Χαίρομαι που είναι τόσο ευαισθητοποιημένος όσον αφορά τις προτεραιότητες μας ο εισηγητής. Κάτι που δεν μου αφήνει πολλά να πω. Απλά θα αναφερθώ σε ένα θέμα ε, ισχυρίζεστε ότι η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για το Συμβούλιο και για την Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό που εγώ δεν βλέπω είναι την ανάγκη να μαχηθούμε για την ασφάλεια της Ευρώπης ε, καταπολεμώντας την παραπληροφόρηση όσον αφορά την Ευρώπη. Εδώ αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή τηλεόραση, στην πρόθεση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, ε τα βλέπουμε αυτά στην έκθεση, αλλά η ευρωπαϊκή ασφάλεια ε, καταπολεμά επίσης και την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση. τις ε, πύλες μέσω των οποίων στρατολογούνται ε, μαχητές στη Συρία. Είχαμε μια γνωμοδότηση εδώ και είναι κατέστη ότι πρέπει να βρούμε πόρους για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χέλγα Τρούπη. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το γενικό στόχο της Κομισιόν. Ανάπτυξη, απασχόληση και ασφάλεια. Και ξέρετε, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, τον οικολογικό μετασχηματισμό επίσης, ε, μια κοινωνία για όλους. Μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε ένα καλό μέλλον για την Ευρώπη χωρίς τη σωστή παιδεία, ε, συμμετοχή στα πολιτιστικά ε, δεν πρόκειται να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση όπως τη θέλουμε. Ε, δεν μπορούμε να λειτουργούμε μονομερώς. Πρέπει να βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα. Και κάτι άλλο, απλά να το αναφέρω, όχι να το επαναλάβω, θεωρώ ότι πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό του Erasmus Plus αντί να βγάζουμε τα χρήματα από το Erasmus Plus και να τα στέλνουμε σε άλλες νέες ιδέες, ακόμη και αν είναι καλές. Αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε για τον προπολογισμό του 2018, σαφώς, και ειδικότερα για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες. Για να πετύχει κανείς στόχους, Όπω είπα, δηλαδή, να έχουμε μια πιο ανοιχτή κοινωνία, περισσότερες ευκαιρίες για μετανάστες και πρόσφυγες και μειονεκτούς ομάδες και τους νέους. Για να γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον τομέα αυτών. Θα ήθελα να επισημάνω δύο άλλα σημεία, τα οποία είναι σημαντικά για εμά. Η ε, σωστή ε, η δημοσιονομική διαχείριση του βραβείου ε, Λάξ ε, που δείχνει ποιο είναι το ευρωπαϊκό αφήγημα στους ευρωπαίους πολίτες, πώς συμμετέχουν οι πολίτες, ε, πώς τους παρέχεται μια δυνατότητα να ε, βλέπουν ευρωπαϊκές κινηματογραφικές παραγωγές στη γλώσσα τους. Και φέτος θα ανοίξει ο Ευρωπαϊκός Οίκος Ιστορίας και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο προπλογισμός εκεί είναι ο σωστός. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν όταν θα δώσουμε την γνωμοδότησή μας για το Γενικό Εισηγητή του Προπολογισμού το 2018. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για αυτές τις δύο τελευταίες ε, επισημάνσεις για τον Νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και το βραβείο Λουξ. Το μουσείο θα, ξεκινήσει, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε, να το επισκεφθούμε. Δεν ήταν έτοιμο ακόμα. Ήμουν μάλλον επιφυλακτική, αλλά αρχικά τουλάχιστον. Πρέπει όμως να σας πω ότι ε, πράγματι φαίνεται ως ένα πολύ θετικό μέσο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την επαρκή χρηματοδότηση ώστε να μπορεί πράγματι το, όχι μόνο η έναρξη να στεφθεί με επιτυχία, αλλά και η λειτουργία του μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Φίμαϊρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε το λόγο? Όχι. Κύριε Μουρεσάν, τότε ε, ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ συνάδελφοι για όλα όσα μας μου είπατε για το Euronews, για το βραβείο Lux, για το Euronet, για, τον, ε, για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Τα έλαβα υπόψη. Το Εράσμους αποτέλεσε μια από τις προτεραιότητες μου από την αρχή. Βλέπετε ότι κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω δημοσίω για τον προπολογισμό, το αναφέρω. Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι πρόκειται για μια καλή επένδυση. Όχι μόνο εξοπλίζει τους νέους ανθρώπους με περισσότερες γνώσεις ε, για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ε, όχι μόνο με εξάσκηση των γλωσσών που μαθαίνουν στο σχολείο και στα πανεπιστήμια, τους εξοπλίζει όπως είπα και με εμπειρία απαραίτητη για να βρει κανεί ε, δουλειά με περισσότερες γνώσεις για την Ευρώπη τους καθιστά λιγότερο ευάλωτους ενώπιον του λαϊκισμού. Πιστεύω λοιπόν ακράδο ότι πρόκειται μια εξαιρετική επένδυση και αποτελεί μια από τις βασικές μου προτεραιότητες. Ε, να ε, δω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σας ε, και στη δική μας συνεργασία κατά τη διάρκεια του έτου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Δεν θα είναι εύκολο βεβαίω, αφού και εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβετε υπόψη σα διάφορα συμφέροντα, διάφορε απόψει σας εύχομαι σε κάθε περίπτωση κάθε επιτυχία στο έργο σας και προσβλέπω στην καλή συνεργασία και με τη δική μας επιτροπή. Λοιπόν, συνάδελφοι, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της συνεδρίασής μας. Κοιτώ την ε, αποδεκατισμένη μας ε, αίθουσα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν θέματα για τα διάφορα, οπότε το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, 4 Μαΐου, 9 έως 12, 12.30 και από 3 το απόγευμα έως 6.30 το απόγευμα το βράδυ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς. Α, η Χέλγα θέλει να πει κάτι. Έχω ένα ερώτημα για την ε, ε, ημερήσια διάταξη για, το, για την 1η Μαΐου. Ε, για, την, ε, ε, για τα εγγένεια. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ε, του, του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ε, θα προσπαθήσω να ακυρώσουμε το, έργο μας ε, για, την ε, απογευματινή συνεδρίαση για να μπορέσουμε να πάμε στα εγγένεια αυτά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε γιατί νομίζω ότι τελειώσαμε πάρα όλα τα θέματα τη σημερινή συνεδρίαση, τα οποία φοβόμουν ότι θα πρέπει να τα μεταφέρουμε στην επόμενη συνεδρία Από αυτή την άποψη, ε, το πιο πιθανό είναι ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ελεύθερο το απόγευμα εκείνη τη ημέρα για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και στα, στα εγγένεια του οίκου τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλου για την παρουσία σα, του Δερβινή και εύχομαι.